εξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και θέλω πρώτα να παρακαλέσω να πάρει το λόγο η εισηγήτρια, η κυρία Μαριέλ Γκαλό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πόσο η νομική είναι ακριβής, καμιά φορά ανυπόμονη για την επίλυση των νομικών προβλημάτων των δυσκολοτέρων. Και πρέπει να πω ότι στην Επιτροπή Ζουρή, στην Νομική Επιτροπή, ακόμα και η μη νομική είναι ανυπόμονη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διαβουλεύσεις όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 90 δημοσίευσε μια σειρά εγγράφων, ανακοινώσεων, έγγραφα εργασίας που ασχολούνται με το θέμα, τα οποία ακολουθήθηκαν από δημόσιες διαβουλεύσεις. Το Κοινοβούλιο ήδη είχε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό πλαίσιο για τι εταιρείε συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών στα πλαίσια των νοματικών δικαιωμάτων και των διαφόρων συναφών δικαιωμάτων. Στο ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου του 2004 και στο ψήφισμα της 13ης Μαρτίου του 2007 και 25 Σεπτεμβρίου του 2008 Κατά τη διάρκεια τη παρούσης θητείας, το Κοινοβούλιο επανέλαβε το ερώτημά του, έτοιμά του μάλλον, κυρίως το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου του 2011, με τίτλο «Ελευθερώστε το δυναμικό ε, του δημιουργικού και πολιτισμικού τομέα» και μια έκθεση που την έχω υπογράψει εγώ, αναφέρεται στο θέμα, που υιοθετήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2010. Όπως το διευκρινίσατε και στην ανακοίνωσή σας στις 24 Μαΐου του 2011, η μελλοντική πρόταση για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία πραγματικής ενίας αγοράς ψηφιακής. Θα πρέπει πανευρωπαϊκές άδειες ή πολυκρατικές αν θέλετε να υπάρχουν αλλά γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο αυτό. Η επαναμοδοποίηση ε, των τίτλων και των θεμάτων είναι δύσκολο να επιτρέπεται σε, μια σε έναν φορέα να δίνει μια άδεια για μια συνολική ομάδα δημιουργημάτων. Θα πρέπει οι εταιρείε λοιπόν διαχείρισης, συλλογικής διαχείρισης των ε, δικαιωμάτων να εγγυάται την πολιτισμική πολυμορφία τονώνοντας τη δημιουργικότητα, αλλά ξέρουμε τους γλωσσικούς και πολιτισμικούς φραγμούς που υφίστανται. Θα πρέπει τέλος αυτές οι εταιρείε συλλογικής διαχειρίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν την αμοιβή όλων των δημιουργών, τη φροντίδα έως δημιουργούς, από τους διεθνείς στάρ μέχρι και τους πιο άγνωστους ε, δημιουργούς. Στην πρότασή σας λοιπόν, πώς σκοπεύετε να πετύχετε ισορροπία μεταξύ το αναγκαίο εξυγχρονισμού της συλλογική διαχείρισης από τη μια, κυρίως να καλύπτονται όλες οι χρήσεις στο διαδίκτυο, αυτό από τη μια λοιπόν, και από την άλλη πώς εξισορροπείται αυτό με την προστασία και την αμοιβή των δημιουργών και ε, να προστατεύεται και η δημιουργική πολυμορφία ταυτόχρονα. Και τελευταίο ερώτημα κύριε Επίτροπε, θα το περιμένετε σαν ερώτημα βεβαίως, σε ποια προθεσμία θα μας προτείνετε, σε πόσο χρόνο θα μας προτείνετε ένα τέτοιο κείμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci, Madame Gallo. Commissaire Barnier, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την Μεριέλ Ελγκάλο εν ονόματι της Επιτροπής που εκπροσωπεί με απασχολεί αυτό το θέμα για την μελλοντική νομοθετική πρόταση για τα συλλογικά πνευματικά δικαιώματα. Ποιο είναι το δικαιωμένο αυτή η συλλογική διαχείριση να εξυπηρετεί την ενιαία αγορά ε, την εποχή του διαδικτύου. Να ε, ζήσουν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, να εφαρμόζονται ε, σε πιο σφαιρικό επίπεδο. Τη σημερινή εποχή, του σημερινούς καιρούς Κυρία Καλό, ξέρετε ότι τώρα η εποχή του διαδικτύου, την εποχή αυτή την ευρωπαϊκή είναι περίπλοκο το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, αφορά την προστασία δικαιωμάτων και online και offline. Όχι μόνο όσον αφορά τους δημιουργούς, αλλά όσον αφορά τους καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή εκτελεστές, ε, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς, ε, τους εκδότες, ακόμα και τους ε, διαφωνικούς σταθμούς. Έχουμε Έχουμε μεγάλες εταιρείες διαχείρισης όπως αυτή που προστα... η εταιρεία που προστατεύει τους δημιουργούς αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης και τις εταιρείε που εισπράττουν τις αμοιβέ που συνδέονται με την αντιγραφή και τα... την αναπαραγωγή. Αν ασχοληθούμε με τη συλλογική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αυτή καθεαυτή είναι ένας τομέας ε, της τάξης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη και μόνο 4,6 δις ευρώ αντιπροσωπεύει ε, συμπεριλαμβάνοντας περίπου καμία εκατοστή διαχείριση από αυτές τις εταιρείε. Αυτή η συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι περίπλοκο διότι έχουμε καμία εκατοστή της εταιρείας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ε, που βρίσκονται στα διάφορα κράτη-μέλη και συμμετέχουν ενεργά στην πολιτισμική ποικιλομορφία σε κάθε κράτος και αυτές όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν δεόντως στο διαδίκτυο και στη ζήτηση που καλύπτει πάρα πολλές χώρες και αναπτύσσεται. Αυτή η συλλογική διαχείριση θα πρέπει να εξυπηρετεί και τους δικαιούχους και τους χρήστες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σήμερα αυτή η συλλογική διαχείριση να ε, εξυπηρετεί εξίσου και την ενιαία αγορά. Η προσφυγή συλλογική διαχείριση πάνω απ' όλα είναι ένα θελοντικό διάβημα και είναι επιλογή που πολύ συχνά επιλέγουν οι δημιουργοί. Επιτρέπει την απόκτηση της αδείας από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών και για μια κάλυψη δικαιωμάτων που είναι η πιο εκτεταμένη δυνατή θα πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των δικαιούχων και να εξασφαλίζει την αμοιβή όχι μόνο, όπως είπατε κύριε Γκαλό, εκείνων που είναι οι πλέον γνωστοί, η στάρ, αλλά να καλύπτει εκείνους και εκείνες που είναι λιγότερο γνωστοί και που έχουν δικαίωμα στην ίδια προστασία. Ιδού δύσκολο να εξευρεθούν αυτές οι ισορροπίες. Το θέμα συλλογική διαχείρισης διαιρεί πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι θέσεις και οι γνώμες ε, είναι πολλές φορές αποκλίνουσες. Παράλληλα, η αγορά εξελίσσεται τάχιστα. Οι χθεσινέ ανάγκες δεν είναι πλέον οι σημερινέ ανάγκες. Κυρίε και κύριοι, υπενθυμίζοντα τον περίπλοκο χαρακτήρα του θέματος και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξηγούν εν μέρη κυρία Γκαλό το χρόνο που χρειάζομαι ούτως ώστε με κάθε σοβαρότητα, με κάθε επίγνωση να επεξεργαστώ αυτή την ε, πρόταση τούτου λεχθέντος να πω κάποια πράγματα για τη μελλοντική πρόταση οδηγίας. Στην ανακοίνωσή μας που υπενθυμίσατε της 20 Μαΐου του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να καλύψει όχι μόνο τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων που καλύπτουν τη μουσική online, αλλά δημιουργεί και μια βάση κοινών κανόνων για όλε τι εταιρείε συλλογική διαχείριση, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα που ασκούν. Αυτή η απόφαση έγινε καλώ δεκτή, κυρίω στα κράτη-μέλη. Ε, έκτοτε εργαζόμεθα με αυτό το στόχο διευρύνοντας το πεδίο που θα καλύπτει η μελλοντική μας πρόταση. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, εξέφρασαν την άποψή τους μέσω διαβουλεύσεως. Αυτές οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί σήμερα. Ε, έκανα χωρίς αυτοσχεδιασμό, το επαναλαμβάνω, σοβαρά, ακούγοντας όλους. Και γι' αυτό, εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα είμαι σε θέση να παρουσιάσω Κατά τη διάρκεια της άνοιξης που έρχεται θα υποβάλω αυτή την πρώτη οδηγία μια και μου ζητήσατε κάποιο χρονικό διάστημα για να προχωρήσω περισσότερο εφόσον έχω την ευκαιρία και να αναφέρω κάποια πράγματα, να μπω σε λεπτομέρειες. Ζητώ από τις υπηρεσίες μου να επεξεργαστούν αυτή την πρόταση ε, που εμπεριέχει δύο πτυχές ε, βασικές. Πρώτα απ' όλα θέλουμε οριζόντιους κανόνες διαφανείας και διακυβερνήσεως. Αυτή η πρώτη οριζόντια πτυχή αφορά εναρμονισμένους κανόνες για και διαφανείας εφαρμοστέους ε, σε όλε τι εταιρείε συλλογική διαχείριση στην Ευρώπη. Αυτοί οι κανόνε θα πρέπει να δημιουργούν ισότιμε συνθήκε για όλε τι εταιρείε και θα βελτιωθεί η λειτουργία τους προς όφελος όλων των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των υπηκών άλλων κρατών μελών. Δεν μπορούμε να μελήσουμε μάλιστα ότι κάθε εταιρεία συλλογική διαχείριση στην επικράτειά τη χειρίζεται τα δικαιώματα που συνδέονται με τη μετάδοση. Όχι ραδιοφωνική, όχι μόνο των μελών, αλλά και των μελών εταιριών διαχείριση ε, εταιριών του εξωτερικού. Αυτή λοιπόν είναι οριζόντια πτυχή α, ε, της μελλοντική μας α, ε, προτάσεως. Δεύτερη πτυχή που περιέχει ειδικοί κανόνες όσον αφορά την μουσική στο διαδίκτυο, online που θα συνδέεται με τι εταιρείε που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική online, εξασφαλίζοντα υψηλό επίπεδο διαφάνεια και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και προ του δημιουργού και προ του χρήστε, θέλουμε να προτείνουμε ένα σαφέ νομικό πλαίσιο προ διευκόλυνση τη παροχή από τι εταιρείε διαχείριση των αδειών που καλύπτουν πολλέ επικράτειε για τη μουσική online. Αυτέ οι άδειε θα ευνοήσουν την επανομοδοποίηση των διαφόρων ε, ε, έργων ε, και θα καθορίζει και τον αριθμό των αναγκαίων αδειών. Θα λάβουμε υπόψη στο βαθμό του δυνατού σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσέγγιση μα στη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματά του και έγγραφα εργασία. Αυτά ήθελα να σα πω ότι προσωπικά και οι ομάδε μου και εγώ προσωπικά επεξεργάζομαι το θέμα. Ο χρόνο που πέρασε, που σα φάνηκε μακρύ, ήταν χρήσιμο για να καταλήξουμε σε στέρεο και ισορροπημένο καλό κείμενο. Είμαι πεπισμένο ότι η πρότασή μα θα συμβάλλει στην επιτάχυνση τη δημιουργία τη ενιαία ψυχιακή αγορά που χρειάζονται και το νομοθετικό πλαίσιο αυτέ οι συλλογικέ εταιρείε διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων με σαφεί κανόνε που θα αναρμονίζουν τι βασικέ αρχέ που αφορούν τη λειτουργία του. Στον τομέα τη μουσική online, η δημιουργία θα βλέπουν να χρησιμοποιούνται περισσότερο τα έργα τους και έτσι και οι πολίτες, και κυρίως οι νέοι, να μπορούν να έχουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και ενωτόμων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Βάσει αυτών των δύο πτυχών που ανέφερα, βέβαια το σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει πρώτα να εγκρίνει το κείμενο και σας είπα τις επόμενες εβδομάδες θα σας το υποβάλουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ και την ερώτησή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα στου ε, ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και θέλω πρώτα να παρακαλέσω την κυρία Μακοβέη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ε, πρόταση της Κομισιόν να προτείνει μια οδηγία για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και καλωσορίζω επίσης και την ανοιχτή νομοθετική διαδικασία που μόλις περιέγραψε ο Επίτροπος που συμπεριλάμβανε και μία διαβούλευση για να ακουθούν οι φωνές των ενδιαφερομένων. Η σύσταση του 2005 της ε, Κομισιόν ε, δεν ρυθμίζει επαρκώς τη συλλογική διασυνορική διαχείριση δικαιωμάτων και τις ε, υπηρεσίες του διαδικτύου. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των δημιουργών στην Ευρώπη και να υπάρξει πολιτιστική ποικιλομορφία σε ένα πλαίσιο νόμιμο και με διαφανή ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα νομικής αβεβαιότητας για τους κατόχους των δικαιωμάτων, για τους χρήστες και ειδικά για τους ε, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν νομική αβεβαιότητα όσον αφορά το ποιο καθεστώς αδειοδότησης ισχύει για τις υπηρεσίες τους θεωρώ πως η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κάποιες από τις εξής αρχές. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε διαχειριστή συλλογικών δικαιωμάτων για τα δικαιώματά τους online σε νόμιμες υπηρεσίες ανεξαρτήτως του που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κάτοχος ή ο διαχειριστής των δικαιωμάτων εντός της Ένωσης. Δεύτερον, δικαιώματα τα οποία συλλέγονται από εταιρείε συλλογική διαχείρισης για λογαριασμό των κατόχων θα πρέπει να διανέμονται δίκαια και χωρίς ε, διάκριση με βάση την κατοικία, εθνικότητα ή εάν είναι συνθέτες, ε, ερμηνευτές ε, ή άλλη κατηγορία κατόχων δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εμπορικούς χρήστες να έχουν πανευρωπαϊκές και πολυταφικές άδειε για το διαδίκτυο και για τα κινητά τηλέφωνα με όρους δίκαιους και χωρίς διάκριση μεταξύ των χρηστών. Και τέλος, σε περίπτωση διαφωνιών θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε μηχανισμό αποτελεσματικό και φτηνό επίλυσης διαφορών, ο οποίος δεν θα περιέχει παράλογο νομικό κόστος. Παρακαλώ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, στην Ευρώπη η ανάπτυξη είναι μια ανάγκη που δεν μπορεί να αναβληθεί πλέον και αυτή εξαρτάται και από τα μέτρα της ε, απελευθέρωσης όσον αφορά τα εμπόδια και τα προνόμια που αφορούν τη εσωτερική αγορά, την ψηφιακή. Και μεταξύ αυτών υπάρχει και ανάγκη για νέα ε, προστασία του copyright, των πνευματικών δικαιωμάτων, κυρίως και του collective rights management, συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Το copyright είναι το 7% του ΑΕΠ της Ευρώπης μας είναι επίγουσα η ανάγκη μεταρρύθμισης. Την περιμένουμε από καιρού. Επανειλημμένα ανακοινώθηκε με προθεσμίε, συγκεκριμένε ημερομηνίε και πρέπει να πω ότι αυτέ οι προθεσμίε και ημερομηνίε δεν είναι σεβαστέ. Εσεί εμέσω το παραδεχτήκατε. Εδώ και δύο χρόνια, πάνω από δύο χρόνια αναμένεται αυτή η οδηγία. Αναμένεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό τη οδηγία 48. Μάλλον τη 29 που είχε καθεστώς εξαιρέσεων ε, ελπίζαμε αυτή η θητεία να είναι η θητεία που θα δημιουργήσει στο πλαίσιο, αλλά σήμερα ε, ακούστηκαν διάφορες ιδεολογικά επιχειρήματα που στερούν τελικά την ελεύθερη πρόσβαση των καλλιτεχνών ε, στο διαδίκτυο και παραλύει αυτή η προσέγγιση. Ε, χρειάζονται νέες τεχνολογικές και νομικές ιδέες για να υπάρχει νέο δικαίωμα πνευματικό που ξεκινά από τη διαχείριση. Υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφέρουσες εμπειρίες και πειράματα, ε, όμως με τις άδειες, τα διπλώματα είχατε κάποια επιτυχία και συγχαρητήρια και σας εκτιμώ. Σε αυτό το θέμα όμως καθυστερείτε. Γιατί αναφερθήκατε και η κυρία Σιγήτη, κυρία Γκαλό, αναφερθήκατε στι δυσκολίε. Πράγματι, υπάρχουν δυσκολίε. Είπατε εν μέρει ότι αυτό δικαιολογεί την καθυστέρηση. Στα λόγια σας διαβάζει κανείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι διαχείρισης και οι δισκογραφική ήχοι ε, εκπροσωπούν μεγάλα συμφέροντα και προστατεύουν το πεδίο τους, το χωράφι τους. Αυτό είναι το βασικό εμπόδιο όχι σε αυτή την εδαφική προστασία, όχι σε υπερβολές παράλογες, όχι σε εκτεταμένες συλλογικέ άδειε, όχι προς νέα μοντέλα επιχείρησης. Ε, λένε ότι θέλουν διαλειτουργικότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, εδώ είναι η ουσία της καθυστέρησης. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν καλά και να μην δημιουργούνται ολιγοπόλια που στρεβλώνουν την αγορά ως και είναι κατά των μικρών εταιριών και πνίγουν τον ε, πνευματικό πλούτο της Ευρώπης και αυτό ζητούμε αυτή την άνοιξη ε, να έρθει επιτέλους αυτή η οδηγία. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπελικουέρ. Ε, η κυρία Βίξτρεμ παρακαλώ από την ομάδα των φιλελευθέρων για δύο λεπτά. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το μικρόφωνο μου. Α, με ακούτε εσείς. Ωραία. Γυρίστε το χρόνο στο μηδέν, παρακαλώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το μέσο μιας ε, τεχνολογικής επανάστασης η οποία είναι πάρα πολύ θετική για τον Ευρωπαίο πολίτη διαδίκτυο σημαίνει απεριόριστη πρόσβαση σε μουσική, βιβλία κτλ. λοιπά Και ακόμα... Κοιτάξτε, αν σκεφτεί κανείς ε, το πώς μεγάλωσα εγώ σε ένα χωριό της Βόρειας Σουηδίας, σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει τελείως. Έχει την ίδια πρόσβαση στα πνευματικά έργα που έχει κάποιος που βρίσκεται στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Πρέπει βεβαίω να υπάρχουν τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι νέοι καιροί σημαίνουν πως τα παλιά συστήματα πρέπει να απλοποιηθούν και να εξυγχρονιστούν. Ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν είναι η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων που θα πρέπει να προσαρμοστεί στον 21ο αιώνα. οι εταιρείε οι οποίες θα διαχειρίζονται τα συλλογικά δικαιώματα για αύριο θα πρέπει να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί βεβαίως μια μικρή επιχείρηση να λειτουργεί σε 27 κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος για να μπορέσει να προσφέρει ένα ε, πανευρωπαϊκό ρεπερτόριο. Θα πρέπει λοιπόν να διαλυθούν τα εμπόδια και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει λοιπόν αυτή η αγορά και αυτό το οποίο προσπαθούμε συνήθως και αυτή είναι η συνήθεια είναι να μένουμε σε αυτό το οποίο έχουμε αντί να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Έτσι ερμηνεύω εγώ την βραδιπορία της ε, Κομισιόν στο θέμα αυτό. Η Ευρώπη χρειάζεται πολιτική ηγεσία, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει πως μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, αναμένω από εσά περισσότερα. Και να σας πω πως εγώ και η ομάδα μου θα συνεισφέρουμε επικοδομητικά σε αυτό για να έχουμε μια πρόταση η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στην ψηφιακή αγορά και θα λειτουργεί μια πρόταση του 21ου αιώνα. Πέσω την κυρία Λίχτεμπεργκερ από την ομάδα των Πρασίνων. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Εκπλήσωμε για το ότι πάλι ανακοινώνεται αναβολή του φακέλου αυτού γιατί προξενεί έκπληξη το ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Από το 2005 συζητάμε το θέμα αυτό. Από το 2005 υπάρχει και η σύσταση της Κομισιόν η οποία ε, έχει οδηγήσει και σε προβλήματα στην αγορά αυτή τη στιγμή και πιέζονται πάρα πολύ οι μικροί διαχειριστές δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε αυτή την πρόταση και τη χρειαζόμαστε κατεπηγόντως. Γιατί πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της εδαφικότητας. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ο κόσμος αλλάζει, δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα. Δεν είναι πλέον μικρές οι διασυνοριακές συνταλλαγές. Επίσης, κατεπήγον είναι πως οι καταναλωτές θα πρέπει να ενισχυθούν και εντός της ε, κοινωνίας τους. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά σε κάποια από αυτά η κατάσταση είναι δραματική επίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησε όλα τα θέματα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση της Κομισιόν. Επίσης είναι επίγον ζήτημα γιατί υπάρξει υπάρχει μια παγκόσμια συγκέντρωση στα χέρια αμερικανικών γιγάντιων εταιριών. Ο χρόνος άρα αυτή τη στιγμή ευνοεί τους δεινόσαυρους της αγοράς και όχι ε, αυτό το οποίο χρειάζεται για να ζήσει η ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, μια άλλη κουλτούρα δηλαδή πέρα από το mainstream, η οποία θα επαναγωνιμοποιήσει μετά ακριβώς αυτό το mainstream. Δεν θέλετε όμως να πάτε σε μια γρήγορη διαδικασία, κύριε Επίτροπε. Καμένους ομιλητές και θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Φρανσουάζ Καστέξ, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με τις προλαλήσατες ότι πρέπει να διεκπαιρεωθεί γρήγορα αυτό το ζήτημα των εταιρεών συλλογική διαχείριση και συμφωνώ με την πρόταση που διατυπώσατε, δηλαδή για την εναρμόνιση των οριζόντιων κανόνων σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και σε ό,τι αφορά την, ε, τις μουσικές επιγραμμικές υπηρεσίες. Να τονίσω και το στόχο ε, της δίκης αμοιβή για τους καλλιτέχνες. Εδώ και κάποια χρόνια το ζήτημα των αποδοχών των καλλιτεχνών αναφερόταν παρά μόνο σε ό,τι αφορούσε παραβιάσεις ε, δικαιωμάτων πραγματικής ε, ιδιοκτησίας και η χρήση του διαδικτύου ήταν ο ποντιπομπέος τράγος για κάποιες απώλειες εσόδων. Στα site όμως ε, των επιγραμμικών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο λαμβάνουν οι καλλιτέχνες. Γι' αυτό θα πρέπει αυτό το θέμα των αποδοχών των καλλιτεχνών να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Φυσικά και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου των Εταιριών ε, Διαχείρισης ε, στη Γαλλία πέρυσι δημοσίευσε μία έκθεση με καταιγιστικά στοιχεία η οποία επίσης κατήγγειλε ότι υπήρχαν ε, τιμολογήσεις και κρατήσεις για έξοδα το θέμα είναι να μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντό μα ο καλλιτέχνη. Υπάρχουν διάφορες ε, πολιτικές τάσεις, όλες όμως καταγγέλουν το σύστημα που τελικά δίνει μεγαλύτερη σημασία στους ε, μεσάζοντες και όχι στους καλλιτέχνες. Το είπε και η Νίλη Κρούς. Υπάρχει δε ένα αδιαφανές ε, σύστημα που είπε και ο Υπουργός, Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού ότι ουσιαστικά παρακρατά και πολλά από τα έσοδα. Πρέπει να ρυθμίσουμε λοιπόν τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, αλλά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προστασία τους πρέπει να είναι και στόχος μας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις ε, αλλά κυρίως ε, οι χρήστες θα πρέπει να σεβαστούν αυτά τα δικαιώματα των δημιουργών. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω τρεις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και πρώτα θέλω, ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Ζαμπόρσκα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι αντιδράσεις Τη κοινό στην άκτα μας δείχνει πως πρέπει να δημιουργηθεί μια τάξη στην ε, κατάσταση αυτή και είναι άρα πάρα πολύ σημαντικό να ισχύουν οι ίδιες αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναμένω λοιπόν ε, οι κάποιες πρακτικές που ακολουθούνται από κάποιους οργανισμούς συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων να σταματήσουν. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και σε αυτές να οδηγηθούμε όσον αφορά τον καταμερισμό των εσόδων. Θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα η νομοθεσία να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Το θέμα είναι, ε, ούτως άλλο, το θέμα είναι επίσης και ο διαμοιρασμός για ε, μερικά λεπτά. Και αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. România sunt organizate și funcționează cu avizul ORDA un număr de 12 organisme. Ευχαριστώ πολύ. 12 φορείς διαχείρισης, συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, εκ των οποίων 5 ασχολούνται με πνευματικά δικαιώματα και 7 στα διάφορα παρεμφερή δικαιώματα. Τα ποσά μοιράζονται σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν λάβει οι φορεί αυτοί από του ε, χρήστε και με άλλα κριτήρια. Υπάρχουν κοινά ταμεία, υπάρχουν κριτήρια ειδικά. Ανάμεσα στο 2004 και 2009 το ποσό που συλλέχθηκε από αυτέ τι ε, φορεί ε, ε, πολλαπλασιάστηκε επί πέντε. Αυτή είναι σημαντική πρόοδο και αυτό δείχνει ότι οι δικαιούχοι, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων γνωρίζουν ε, τα δικαιώματά του και τα ωφέλη μπορούν να αποκομίσουν όταν μπορούν να προσχωρήσουν σε μια εταιρεία στο διαχείριση. Σα ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια μέτρα προβλέπετε μέσω τη νομοθετική σας πρόταση, ώστε να εγγυάσετε την πρόσβαση των δικαιούχων ε, αυτών δικαιωμάτων, κυρίως των πλέον αγνώστων καλλιτεχνών, σε εταιρείε συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή άδεια και τι θα κάνετε για να υπάρχει μια πρόσβαση των έργων ε, σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είτε μιλάμε τώρα για διάφορα πόρταλ που κάνουν streaming είτε άλλες ε, σελίδες ε, υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες αγορές. Γι' αυτό δεν έχει εξαντληθεί νομίζω το δυναμικό που υπάρχει. Σε σύγκριση δε με τις ΗΠΑ ή την ε, Ασία υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερες δυνατότητες, ειδικά για νέους καλλιτέχνες και που δεν είναι τόσο διάσημοι, δίνει το διαδίκτυο την δυνατότητα να φτάσουν σε ένα μεγάλο κοινό. Και αυτό το οποίο χρειάζεται για να εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό είναι να δημιουργήσουμε το σωστό νομικό πλαίσιο επίση για τις άδειε, γιατί θα πρέπει βεβαίω να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματά τους η δημιουργοί. βεβαιω η Ευρώπη δεν έχει μόνο ιστορικό ρόλο να παίξει στον πολιτισμό, θα πρέπει ε, στοχευμένο να δούμε τι θα κάνουμε στο ψηφιακό πεδίο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, βουλευτές για τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα. Όλα τα σημείωσα και θα τα λάβω υπόψη. Ολοκληρώνοντας ε, το προπαρασκευαστικό έργο μου, τις διαβουλεύσεις που έχω, θέλω να πω, όπως είπα και στην κυρία Γκάλο και στην πρώτη μου απάντηση, για ένα τέτοιο θέμα τόσο σοβαρό, που φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και διάφορα ε, συμφέροντα που υπάρχουν. Πρέπει όμως να λέμε πως και την νομική πολυπλοκότητα. Ο χρόνος ε, που χρησιμοποίησαμε και που θα ήταν θα, καλό κατά να πούμε συντομότερος, αλλά ήταν απαραίτητος ο χρόνος αυτός για να έχουμε ένα δυναμικό και ευφυές κείμενο. Κυρία Καλό, στο πρώτο της ερώτημα θέτει ένα ζήτημα το οποίο και άλλοι ευρωβουλευτές μου θέσατε, δηλαδή πώς θα εγγυηθούμε στο πλαίσιο αυτής της πρότασης μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δημιουργών αφενός και της πολυπολιτισμικής ε, πολιτισμικότητας και την πρόσβαση των δημιουργημάτων στον περισσότερο δυνατό κόσμο και εξυγχρονισμό της συλλογικής διαχείρισης αφετέρου. Πώ θα τα συμφιλιώσουμε όλα αυτά. Θέλω να σα υπενθυμίσω, αγαπητοί βουλευτέ, ότι η συλλογική διαχείριση είναι ένα ε, ε, πολύ σημαντικό παράγοντα. Είναι μεσάζονται μεσολαβητέ μεταξύ δημιουργού και κοινού. Για το δημιουργό δεν είναι υποχρέωση να περάσει μέσω των εταιριών αυτών συλλογική διαχείριση. Και το λέω κυρίω προ την κυρία Ζαμπόρσκα. Είναι, είναι επιλογή, οικειοθελή του καλλιτέχνη έχει σίγουρα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και όπως είπατε και εσείς κύριε και άλλοι πρόκειται για ένα καθήκον δύσκολο τη στιγμή που οι οργανισμοί αυτοί κάνουν σημαντικές επενδύσεις για τις ε, διάφορες πολυκατοικές αντιδοτήσει και θα πρέπει και τα τεχνικά οικονομικά εμπόδια να τα έχουμε υπόψη μας σε μια αγορά που είναι ακόμη εύθραυστη και αναπτύσσεται ακόμη. Δεν είναι εύκολο για όλους να αναπτύξουν αυτά τα δικαιώματα και τις αδειοδοτήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους ε, δημιουργούς αυτούς εκτός της ψηφιακής εποχής εξού και προτείνω μέτρα τα οποία θα έπρεπε ουσιαστικά να μπορούν να μας κάνουν να επιλέξουμε την καλύτερη δυνατή ε, διασυνοριακή αδειοδότηση. κυρία Καστέξ, κυρία Μερζή, μίλησαν για την ανάγκη καλύτερης διακυβέρνησης και ανέφεραν συγκεκριμένα παραδείγματα που πραγματικά προκαλούν ε, ένα διάλογο, μια συζήτηση και κάποιες περιπτώσεις σίγουρα είναι μη φυσιολογικές. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να είναι καλύτερη διακυβέρνηση. Εμείς έχουμε ενθαρρύνει και ευνοήσει την ε, συνέχιση των δραστηριοτήτων όλων των οργανισμών και εταιριών υπό καλύτερε συνθήκε. Αλλά όπω και εσεί, έτσι και εγώ, πιστεύω ότι οι προτάσει μα θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση τη διακυβέρνηση. Πράγματι, ε, εξηγήσατε κάποια πράγματα για την προθεσμία και καταλαβαίνω τι λέτε. Συμφωνώ και εγώ. Απλά σας ζητούμε υπομονή για λίγες ακόμη εβδομάδες μέχρι ότου καταλήξουμε. Όπως και η κυρία Βίξτρομ, ε, ζητήσατε να προσπαθήσουμε να συντομεύσουμε τις προθεσμίε. θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά πρέπει και εσείς να αναγνωρίσετε ότι το χρόνο αυτό τον αξιοποιήσαμε και γενικότερα για στον ευρύτερο κλάδο αυτό τη ιδιοκτησία για να σημειώσουμε πρόοδο και σε άλλα σημαντικά θέματα. Εσεί είπατε για την ευρεσιτεχνία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Μπορώ να σα μιλήσω εγώ για τα ορφανά έργα και τη διαχείρισή τους. Ή για το παρατηρητήριο σε σχέση με τις παραβάσει στον τομέα τη πνευματική ιδιοκτησία που αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα στο ημικύκλιο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση αναθεώρηση τη οδηγία για την εφαρμογή ε, των δικαιωμάτων διανοητική ε, ιδιοκτησία, είναι υποεκπώνηση αυτό το νομοθέτημα τον κύριο Βιτορίνο, συνάδελφό μου πριν από κάποια χρόνια, ε, τον παρακαλέσαμε να γίνει να αναλάβει την ε, εκπόνηση αυτής της πρότασης και τη μελέτη. Επίσης μας ενδιαφέρει και ο οπτικοακουστικός τομέας ε, και θα έχουμε σχετικές εξελίξεις μέχρι το καλοκαίρι. Κύριε Βίξτρο, μεταξύ άλλων και αν κατάλαβα καλά, ανέφερε και το μέλλον των οργανισμών συλλογική διαχείριση μικρή κλίμακα. Πράγματι, δεν είναι όλοι οι οργανισμοί συλλογική διαχείριση το ίδιο ε, μεγάλοι. Το μεγαλύτερο μέρος των εισόδων προέρχονται από άδειες που δίδονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε κανάλια τηλεόρασης, σε παραγωγούς δίσκων κτλ. Οι συλλογικοί οι οργανισμοί διαχείρισης θα συνεχίσουν να εκχωρούν αυτές τις άδειες, αλλά σε ένα πλαίσιο πιο αποτελεσματικό και πιο διάφανο. Και νομίζω ότι όλοι εκτιμούν το ότι θα μπορούν να έχουν την πρόσβαση στην αγορά, στην γλώσσα τους. Και αυτό δεν προτιθέμεθα να το αλλάξουμε. Οι κυρίες Βίξτρομ, Τικάου ανέφεραν και το θέμα των ε, ρεπερτορίων που θα πρέπει να είναι διασυνοριακά διαθέσιμα και αυτό είναι σημαντικό για όλους και κυρίως για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί διαχείρισης ε, δυνατότητες να προτείνουν ε, πολυκρατικές ε, αδειοδοτήσεις, αλλά εμείς θέλουμε όλα τα ρεπερτόρια να είναι διαθέσιμα για αυτές τις άδειε. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Για την κυρία Μακοβέη, που ανέφερε το θέμα του ανταγωνισμού στη λειτουργία των οργανισμών συλλογική διαχείριση, Πράγματι, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία αυτών των οργανισμών και περισσότερες δυνατότητες και για τους δικαιούχου να μπορούν με τα λόγω γνώσεως να κάνουν τις επιλογές τους. Γιατί θα υπάρχει ένα κοινό ε, πλαίσιο και ισότιμοι κανόνε για τη διαχείριση τη συλλογική και του οργανισμού αυτού στην Ευρώπη. Σίγουρα θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να βελτιώσετε αυτό το κείμενο, αλλά νομίζω ότι και οι εμπορικοί χρήστες και οι δικαιούχοι θα μπορούν πλέον ευκολότερα να συγκρίνουν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν οι διάφοροι οργανισμοί συλλογική διαχείρισης. Και έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το δημιουργικό δυναμικό που υπάρχει στην Ευρώπη πιο αποτελεσματικά. Η κυρία Ζαμπόρσκα επίσης ανέφερε τη συμφωνία ΑΚΤΑ. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι απασχολεί πολλούς από εσάς. Το ανέφερα και σε προηγούμενη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το κείμενο και ο συνάδελφος Δεχούχτε τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου ε, θα έρθει σε όλες τις να συμμετέχει για να δούμε με πιο ήρεμο τρόπο, με πιο αντικειμενικό τα θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία άκτα. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν και αυτό το σημείο σας ευχαριστώ που μου θέσατε την προφορική αυτή ερώτηση αλλά και ε, για τα σχόλια που κάνατε στην απόψινή συζήτηση στην πρότασή μας για τη συλλογική διαχείριση των ε, δικαιωμάτων των δημιουργών θα βρείτε όλες αυτές τις σχετικές προτάσεις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον προγραμματισμό των διαθωτικών ταμείων για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση